Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων ε, στη Γουατεμάλα για την τραγωδία που προκλήθηκε από μια περκαγιά η οποία ξέσπασε την περασμένη Τετάρτη σε έναν ε, χώρο για ε, ανηλίκους ε, θύματα βίας στο Σαν Χωσέ Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προκειμένου να γνωρίζουμε τα αίτια του τραγικού γεγονότος και να αποδοθούν και πιθανώς ευθύνες. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι θα έπρεπε να την χάνουν καλύτερης προστασίας. Όπως γνωρίζετε την προηγούμενη εβδομάδα γιορτάσαμε την ημέρα της γυναίκας. Ε, επέμεινα ο εορτασμός αυτός να μην ε, παραμείνει απλώς ε, μια ευκαιρία στη θεωρία, και μέχρι ότου οι γυναίκες ε, συνεχίσουν να είναι θύματα βίας, ε, διακρίσεων, ε, καταναγκαστικών γάμων, αποκλείονται από το χώρο εργασίας και από τις πολιτικές ευθύνες, πρέπει κάθε μέρα του χρόνου να δίνουμε μάχη προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών